Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην κοινή επιτροπή της, ε, κοινή συνεδρία της Επιτροπής ΑΦΕΤ ε, Ελευθεριών ε, Ανάπτυξης. Θέλω να ευχαριστήσω τους αδέλφους που είναι εδώ σήμερα, που κατάφεραν να φτάσουν Δευτέρα μεσημέρι παρά τις δυσκολίες στις μεταφορές. Έγκριση της μίλης διάταξης πρώτα, δεν υπάρχουν σχόλια φαντάζομαι και περνάμε στο σημείο 2, ανακοινώση του Προέδρου. Ούτε εδώ υπάρχει κάτι. Στο σημείο 3, τα πρακτικά που πρέπει να εγκριθούν των προηγούμενων συναντήσεων, 23 Ιανουαρίου, 1 Φεβρουαρίου, εφόσον δεν υπάρχουν σχόλια, εγκρίνονται και τα πρακτικά. Οπότε πάμε ήδη στο σημείο 4 της εμείς διάταξης. Θέλω να καλωσορίσω τη Λουίζ Άρμπορ, όπως ε, θα γνωρίζετε, μιας και έχει έρθει συχνά στο Ρεπέγο Κοινοβούλιο, είναι η ύπατη εκπρόσωπος ε, των Ηνωμένων Εθνών για τη Διεθνή Μετανάστευση. Καλώς ήρθατε. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που είστε εδώ σήμερα. Ως ε, ειδική εκπρόσωπος, η κυρία Άρμπουρ παρακολουθεί τις ε, πτυχές που έχουν κάνει με τη μετανάστευση ε, στη Συνόδο Κορυφής των Ηνωμένων Εθνών και συνεργάζεται με τα κράτη-μέλη ε, για μια σφαιρική αντιμετώπιση της μετανάστευσης. Τη γνωρίζουμε την κυρία Άρμπορ, είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψη μαζί της ε, πολλές φορές στο παρελθόν, πιο πρόσφατα στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, για το Παγκόσμιο Σύμφωνο, για τη μετανάστευση, αλλά και στο παρελθόν ε, ως ε, είπατε εκπρόσωπος των Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Να κάνω ένα σχόλιο από τη δική μας πλευρά ως ε, Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εμείς θεωρούμε ότι είναι σημαντικό τα κοινοβούλια να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο κατά την ανάπτυξη και την εφαρμογή του Παγκόσμιου Συμφώνου παρακολουθούμε τη διαδικασία του Παγκοσμίου Συμφώνου στενά και η σημερινή συζήτηση είναι μία από πολλές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο Κοινοβούλιο αυτό γύρω από το ζήτημα αυτό. Έχουμε εμπλακεί εντατικά και έχουμε και εμπλέξει και πολλούς άλλους φορείς ε, από τα Ηνωμένα Έθνη και άλλες διεθνείς οργανώσεις ε, καθώς και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα τελευταίο σχόλιο μια, ένα ψήφισμα της Ολομέλειας για το Παγκόσμιο Σύμφωνο ε, είναι υπό προπαρασκευή και θα εγκριθεί στην Ολομέλεια του Απριλίου μετά από συζήτηση με την κυρία Μογκερίνη, την είπατε εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Ζίμπελ ε, για τα πρώτα σχόλια από την Επιτροπή Ελευθεριών. Ναι, χαίρομαι που είπατε αντιπρόεδρος. Είμαι απλά συντονίστρια όμως στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, λέει η κυρία Ζίπελ. Πάντως ε, ευχαρίστως να προεδρεύσω. Ναι, σας ε, έδωσα μια προαγωγή, λέει ο πρόεδρος, ίσως την επόμενη φορά. Ε, εγώ πραγματικά εκτιμώ που είναι και πάλι εδώ μαζί μας η Λουίζ Άρμπορ και χαίρομαι επίσης που βλέπω συναδέλφους από διάφορες επιτροπές. Ελπίζω λοιπόν να έχουμε μια καλή συζήτηση σήμερα το απόγευμα. Το Κοινοβούλιο μας και η Επιτροπή Ελευθεριών ιδιαιτέρως έχουν δώσει μεγάλη προσοχή σε όλη αυτή τη διαδικασία σε σχέση με το Παγκόσμιο Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών. Αναγνωρίζουμε ότι αυτό αποτελεί μια ιστορική ευκαιρία για να πετύχουμε ε, μια σειρά από δεσμεύσεις, μια σειρά από αρχές που θα διέπουν τα ζητήματα διεθνούς μετανάστευσης. Ήδη το Σεπτέμβριο του 2016 αυτό το, το, το κοινοβούλιο συμμετείχε στην αντιπροσωπεία υπό τη Σεσίλια Βίκστρομ στη Σύνοδο Κορυφής για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες όπου ε, ενεκρίθη η περίφημη δήλωση της Νέας Υόρκης. Μια σειρά από δράσεις λοιπόν έχουν αναλυφθεί για ενεργή συμμετοχή, ενεργή συνεισφορά σε αυτή τη διαδικασία έχουμε ήδη ε, οργανώσει και στο παρελθόν και αναφέρθηκε αυτό συναντήσει με την κυρία Άρμπορ. Ε, συναντήσαμε και τους συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια για το θέμα αυτό σε συνεργασία με την Επιτροπή ΑΦΕΤ και με συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων σε αυτή τη διαδικασία. Γνωρίζουμε ότι το ψήφισμα, το είπε και ο κ. Μακάλιστερ, ε, πρόκειται να ψηφιστεί στην Ολομέλεια του Απριλίου και θα εκφράζει βεβαίως ε, την υποστήριξή μας στις αρχές της δήλωσης της Νέας Υόρκης και ε, στην διαδικασία για τη δημιουργία ε, ενώ μιας σφαιρικής διακυβέρνησης με ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα διεθνής μετανάστευσης. Λυπάμαι όμως για την απόφαση της Αμερικανικής κυβέρνησης να σταματήσει τη συμμετοχή της στις διαπραγματεύσεις για αυτό το παγκόσμιο σύμφωνο. Βεβαίως, ε, ίσως αυτό να είναι και μια ευκαιρία να αναλάβουμε εμείς ε, τα ηνία ως Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτή τη διαδικασία και τα κράτη-μέλη θα πρέπει εδώ να ε, επιδείξουν ενότητα, να μιλήσουν μια φωνή υπέρ ενός ενιαίου διεθνούς καθεστώτος για την διαχείριση της μετανάστευσης. Θα ήθελα να πω τέλος ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει σκοπό να συμμετάσχει στην διάσκεψη που θα οργανωθεί στο Μαρόκο τον Δεκέμβριο. Και η κυρία Άρμπουρ ως ε, γενική γραμματέας για την διακυβερνητική αυτή διάσκεψη θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να εξασφαλίσει ότι η παρουσία μας ε, θα καταστεί εφικτή. Ειλικρινά, πιστεύω ότι το Ελληνικό Κοινοβούλιο θα, μπορού, θα μπορούσε και θα μπορέσει να συνεισφέρει σε αυτή τη συζήτηση λαμβάνοντας υπόψη και τον νομοθετικό μας ρόλο για ζητήματα που σχετίζονται με τη μετανάστευση και το άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα από εκεί και πέρα, ως Επιτροπή ΛΥΜΠΕ ε, θα δώσουμε τώρα το λόγο, αφού ακούσετε την άποψη της ΛΥΜΠΕ, θα δώσουμε το λόγο στις αμέσως στην κυρία Άρμπορ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω τους ε, προέδρους των τριών επιτροπών που μου έδωσαν την ευκαιρία να απευθυνθώ μαζί σας σήμερα ε, σχεδόν στη μέση αυτής της διαδικασίας διαπραγμάτευσης ε, για το Παγκόσμιο Σύμφωνο ε, για μια ασφαλή, συντεταγμένη και νόμιμη μετανάστευση. Έχουμε ολοκληρώσει δύο γύρους από τους έξι γύρους διαπραγματεύσεων. προς την έγκριση του κειμένου αυτού που προβλέπεται τον Ιούλιο όταν λέω έχουμε ολοκληρώσει, δεν, δεν συμπεριλαμβάνω τον εαυτό μου. Το Παγκόσμιο Σύμφωνο είναι μια πρωτοβουλία, μια διαδικασία της των και των κρατών μελών. Ο, μόνιμος εκπρόσωπος της Ελβετίας και του Μεξικού στη Νέα Υόρκη διευκολύνει την όλη διαδικασία και είναι και η βασική υπεύθυνη για το πρώτο σχέδιο κειμένου που ήταν και η βάση της διαπραγμάτευσης έως τώρα. Σε γενικές γραμμές πρέπει να πω ότι κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, ένα έτος ε, εντατικών διαβουλεύσεων, περιφερειακών, θεματικών, είχαμε μια πραγματικά εξαιρετική στάση και συμμετοχή από όλους τους ενδιαφερομένους. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι η μετανάστευση, η κινητικότητα των ανθρώπων γενικότερα παρουσιάζει τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά από περιοχή σε περιοχή του κόσμου. Εδώ μιλάμε για ένα παγκόσμιο σύμφωνο. Είναι πολύ σημαντικό τα κράτη-μέλη, οι διάφορες περιφέρειες να ε, προσέλθουν στις συζητήσεις ε, με ανοιχτό πνεύμα, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά αλλού. Ε, μαθαίνουμε μέσω των παρεμβάσεων των κρατών μελών ότι αντίθετα με διάφορα στερεότυπα τα κράτη-μέλη δεν είναι μόνο κράτη-μέλη προέλευσης ή τράνζιτ ή προορισμού. Ε, τα πιο πολλά, οι πιο πολλές χώρες ε, είναι και τα τρία. Είναι και χώρες προέλευσης και χώρες προορισμού και οι περισσότερες, ε, το μεγαλύτερο μέρος της διεθνής, διεθνούς μετανάστευσης ε, Βεβαίω κινητικότητα αφορά κυρίως το ιστορικό της κάθε χώρα, εδώ μιλάμε για την διεθνή μετανάστευση. Σε μεγάλο βαθμό λοιπόν είναι υποπεριφερειακή, περιφερειακή, υπηρετική και κατόπιν διεθνής. Είναι επικίνδυνο κατά κάποιο τρόπο να μιλήσουμε για κάποια συνένεση σε αυτή την πρώιμη φάση, ε, αλλά μπορώ να πω ότι σε κάποιους τομείς υπάρχει σαφή σύγκληση για να μην πω απόλυτη συνένεση. Θα μπορούσα να πω ότι υπάρχει συνένεση. Ε, Βεβαίω πρόκειται για κάποιους, κάπως γενικά ζητήματα. Στη συνέχεια θα αναφερθώ και στα ε, πιο αμφιλεχόμενα. Θα αναφερθώ και στα ζητήματα όπου πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας. Λοιπόν, είναι σαφές ότι τα κράτη-μέλη έχουν επανεπιβεβαιώσει ότι το Παγκόσμιο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση πρέπει να έχει ως τον άνθρωπο. Δεν είναι μια εμπορική συμφωνία, δεν μιλάμε για ροή κεφαλαίων, μιλάμε για ανθρώπους. Και τα ανθρώπινα δικαιώματα παίζουν ένα κεντρικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. Εξίσου σημαντικό είναι να είναι ότι όλα τα κράτη-μέλη αναφέρθηκαν στη σημασία της εθνικής κυριαρχίας και στο πλαίσιο αυτό υπάρχει αρμοδιότητα αλλά και ευθύνη των κρατών να ελέγχουν τα σύνορά τους και να παίρνουν την απόφαση αυτά για το ποιος εισέρχεται στο έδαφος τους, υπό ποιες προϋποθέσεις. Βεβαίως αυτό υπόκειται στο δίκαιο, στο εθνικό δίκαιο, αλλά και σε κάποιες ε, εδρεωμένες αρχές διεθνούς δικαίου, όπως η αρχή ε, της μη απόκρουσης, της, της μη επαναπροώθησης Εδώ πάντως δεν μιλάμε για κάποιο νομικό δεσμευτικό κείμενο, δεν μιλάμε για κάποια συνθήκη και αυτό μας δίνει ευελιξία. Δίνει ευελιξία στα κράτη-μέλη έτσι ώστε να φτάσουν σε μια, πραγμα... μια, ε, συμφωνία πραγματικής συνεργασίας χωρίς ε, να υπάρχει το άγχος ε, της δέσμευσης γύρω από μια συγκεκριμένη διατύπωση. Παναλάβαμε επαναλάβαμε για άλλη μια φορά, παρότι ευθύς εξ αρχής είχε υποθεί, και σε αυτό το τελευταίο γύρο διαπραγματεύσεων ελέγχθη το πόσο κρίσιμη είναι η σχέση μεταξύ μετανάστευσης και ανάπτυξης. Οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης που είναι το ευρύτερο πλαίσιο εντός του οποίου προχωράει την ατζέντα για την ανάπτυξη του ανάπτυξη των έθνη για πρώτη φορά η μετανάστευση αναγνωρίστηκε ότι παίζει ρόλο στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης ε, ιδιαίτερα στο ότι αφορά στόχο υπαριθμών 10, την ανάγκη μείωση των ανισοτήτων εντό των, χωρών, των κρατών και μεταξύ κρατών. Και τέλος, όπως λέει ε, και το όνομα του όλου εγχειρήματο, μιλάμε για ένα παγκόσμιο σύμφωνο για ασφαλή νόμιμη και συντεταγμένη μετανάστευση. Δεν θέλουμε να προωθήσουμε τη μετανάστευση. Θέλουμε ασφάλεια, θέλουμε μια τάξη, θέλουμε μια νομιμότητα να προσθέσουμε να μειώσουμε την παράτυπη μετανάστευση που συνδυάζεται με πολύ αρνητικές πτυχές ε, για τους ίδιους τους μετανάστες αλλά και για τις χώρες, ε, τις χώρες προέλευσης αλλά κυρίως τις χώρες προορισμού. Έχουμε μάθει πολλά ε, όλοι μαζί σε αυτή τη φάση διαβούλευσης και καθόλου τη διάρκεια των πραγματεύσεων έως τώρα και είναι σημαντικό στην αρχή αυτής της συζήτησης να υπενθυμίσω κάποια πράγματα. Πρώτα απ' όλα το, η κλίμακα της μετανάστευσης σήμερα με βάση την κατανομή του πληθυσμού στην έθνη έχουμε περίπου 250 εκατομμύρια ε, πρόσφυγες, ε, ε, μετανάστες συγγνώμη, Εξ των οποίων ένα ποσοστό είναι πρόσφυγες. Μιλάμε δηλαδή για ανθρώπου που ζουν αλλού από τη χώρα προέλευσή του, από τη χώρα ε, όπου γεννήθηκαν. Αυτό δεν περιλαμβάνει τους ανθρώπους οι οποίοι είναι εν κινήσει, τις ροές δηλαδή, όπως λένε οι, οι πυρογνώμονες. Καλύπτει όμως ε, ε τα αποθέματα των υπάρχοντων μεταναστών. Ε, είναι δύσκολο βεβαίως καθημερινά να μπορούμε να παρακολουθούμε και να μετρούμε ε, τις ροές αυτές. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, αλλά είναι όλο και περισσότερο ένα φαινόμενο μετακίνησης από τον νότο προς τον νότο. Δηλαδή από χώρες του νότου προς χώρες του νότου. Πολύ πιο συχνά από ό,τι προς το βορρά παρά ε, τα όσα ε, μπορεί να, θα μπορούσε να θεωρήσει κάποιος έτσι λοιπόν έχουν πιο, έχουμε πιο κοινά σημεία στις πραγματεύσεις από ό,τι θα μπορούσε να φανταστεί κανείς όταν κατηγοροποιεί τον κόσμο ε, με διαφορετικό τρόπο. Ένα άλλο κρίσιμο ζήτημα που πρέπει να έχουμε κατά νου είναι ότι σε αυτό το τομέα, όπως και σε άλλους, η πραγματικότητα είναι καλύτερη από την αντίληψη που έχουμε. Ορισμένε φορέ ε, δυστυχώς ε, η κοινή γνώμη βασίζεται στην αντίληψη που δημιουργείται και αυτό τελικά διέπει και τις πολιτικές αποφάσει που παίρνονται. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα, είναι διαφορετικά και σε ό,τι αφορά την οικονομική πτυχή. Είναι ένα θετικό φαινόμενο μετανάστευση από οικονομικής πλευράς. Συντριπτικά Αυτές 350 εκατομμύρια, των οποίων 38% είναι γυναίκες, οι γυναίκες μετανάστες ε, ε, εργαζόμενοι που ε, έχουν μεγάλες δυνατότητες απασχόλησης από ότι οι θαγενείς, αυτό οδηγεί στο να στέλνονται χρήματα πίσω στις χώρες προέλευσης, πολύ σημαντικά ποσά, 85% των εσόδων ε, δαπανώνται βεβαίως στη χώρα όπου ζούνε, αλλά το 15% που στέλνουν στην χώρα τους είναι τρεις φορές, ε, τρεις φορές το, συνολικό, το συνολικό ποσό αναψυξιακής βοήθειας. Δηλαδή πρόκειται για φτωχούς ανθρώπους που, που βοηθούν άλλους φτωχούς ανθρώπους, χωρίς να, περνούμε από, χωρίς να περνάνε από επίσημους διάβλους. Ε, είναι μια πραγματική προσπάθεια ουσιαστικά άμεσης επένδυσης στην εκπαίδευση, στο, στην διατροφή αλλά και στη χειραφέτηση συχνά των γυναικών ε, στις τοπικές κοινωνίες. Βεβαίως ε, υπάρχει και ένα κόστος που σχετίζεται συνήθως με την παράτυπη μετανάστευση και αυτό είναι ένα θέμα στο οποίο θα ήθελα να επικεντρωθώ σήμερα. Υπάρχουν ένα-δύο ουσιαστικά ζητήματα που θέλω να αναφέρω. Το πρώτο είναι το ζήτημα αυτό της νόμιμης και της παράτυπης μετανάστευσης. Αυτή η ορολογία έχει πλέον εδρεωθεί είναι καλύτερο από τη ρητορική περί παράνομης μετανάστευσης που τόσο συχνά συνδέεται με την εγκληματικότητα ε, σε ένα, σε πλαίσιο το οποίο δεν αποκρίνεται στην πραγματικότητα. Να αναφερθώ λοιπόν λίγο στο θέμα αυτό της ε, ε, νόμιμης και της παράτυπης μετανάστευσης και θα ήθελα να πω γενικότερα πώς πρέπει να προσεγγίσουμε τα ζητήματα αυτά στο ευρύτερο φάσμα. Ο διαχωρισμός μεταξύ νόμιμη και παράτυπης μετανάστευση μπορεί ε, να χωριστεί σε δύο προσεγγίσεις. Είναι πιο βολικό αυτό. Ε, μπορεί να μην φαίνεται να υπάρχει διαφορά αρχικά, αλλά είναι καλό να υπάρξει διαχωρισμός μεταξύ της νόμιμης μετανάστευσης και των παράτυπων μεταναστών. Η, η παράτυπη μετανάστευση έχει, ουσιαστικά ε, αναφέρεται σε ροές ανθρώπων και όταν μιλάμε για παράτυπη μετανάστευση, σκεφτόμαστε την παράτυπη είσοδο σε μια χώρα και αυτό βεβαίως δημιουργεί αμέσω ε, μια εικόνα περί λαθρεμπορίου, περί εμπορία ανθρώπων, περί μορφ... διαφόρων μορφών εγκληματικότητα που συνδέονται με αυτές τις παράνομες ροέ ανθρώπων, ε, τις παράνομες μετακινήσεις. Όταν όμω μιλάμε για παράτυπου μετανάστε, εδώ μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε μία χώρα, στη χώρα προορισμού τους, είτε χωρίς χαρτιά, είτε, ε, εν σε μία κατάσταση παράτυπη. Υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο, όταν εξετάσουμε ε, ποια πολιτική πρέπει να ακολουθηθεί για να μειωθεί το φαινόμενο αυτό. Θα ήταν τελείως αγαθό να πιστεύει κανείς ότι μπορεί βεβαίως να ε, πάψει να υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Αλλά υπάρχουν πολιτικές που συνεισφέρουν ε, στην αρνητική στάση απέναντι στους μετανάστες και στην εντύπωση που δίνεται ότι οι, με, κυβερνήσεις έχουν χάσει τον έλεγχο των συνόρων και των πολιτών τελικά που ζουν στη χώρα. Ο τελευταίο γύρο διαπραγματεύσεων στη Νέα Υόρκη, όπου τα κράτη-μέλη εκλήθησαν να εξετάσουν τα ζητήματα αυτά, η μεγάλη πλειοψηφία ε, μιλούν για παράτυπου μετανάστε. Θέτουν το θέμα λοιπόν του πώ τα κράτη-μέλη πρέπει να αντιμετωπίσουν τους ανθρώπους που ζουν στο έδαφος τους με, κάποια παράτι, με κάποιον παράτυπο τρόπο. Και εδώ τίθεται το δύσκολο ζήτημα ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υπάρχει μια γενική συνένεση ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, είναι ενιαία, αφορούν όλο τον κόσμο, εφαρμόζονται σε όλους, έχουν να κάνουν με την ίδια την ε, την ανθρώπινη υπόσταση του ανθρώπου και ότι όλοι πρέπει να χαίρουν το δικαιωμάτων αυτών. Ανεξάρτητα από το καθεστώς, του, το μεταναστευτικό του καθενός, ε, αρχίζουν όμως να τίθενται κάποια ερωτήματα. Αυτό που θα πρέπει να συζητηθεί στις διαπραγματεύσεις αυτές είναι πρώτα απ' όλα να υπάρξει μια κάποια σαφήνεια μεταξύ δικαιωμάτων, ε, υπηρεσιών βασικά δικαιώματα, βασικές υπηρεσίες, πρόσβαση σε υπηρεσίες, υποχρεώ, υποχρέωση προσκόμισης κάποιων στοιχείων. Όλη αυτή η ορολογία ε, πιο πολύ δημιουργεί σύγχυση αυτή τη στιγμή παρά διευκρινίζει την κατάσταση. Σε ό,τι αφορά το ποιο είναι ο κοινό παρονομαστή ε, με βάση τον οποίο θα μπορούσαν να συμφωνήσουν τα κράτη-μέλη στα πλαίσια του Παγκόσμιου Συμφώνου. Ακόμα και οι τουρίστε έχουν δικαίωμα σε κάποια μορφή προστασία όταν επισκέπτονται μια χώρα. Και οι μετανάστες, οι παράτυποι, έχουν κάποια δικαιώματα. Κανείς όμως δεν λέει σοβαρά ότι το δικαίωμα ψήφου, παραδείγματος χάρη, θα πρέπει να επεκταθεί σε οποιονδήποτε βρίσκεται στο έδαφος μιας χώρας. Στα πλαίσια λοιπόν των πολιτικών δικαιωμάτων, των ε, κοινωνικών, οικονομικών, πολιτιστικών δικαιωμάτων πρέπει να δούμε ποιες διατάξεις ε, θα πρέπει να πληρώνεται απαρέκλητα από τα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και πού θα υπάρχουν διαχωρισμοί μεταξύ ε, εθνικών, υπηκών, ε, αλλοδαπών, μεταναστών, παράτυπων μεταναστών και τι, ποιες διαφοροποίησεις μπορεί να γίνουν αποδεκτές με βάση το Διεθνές Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Είναι κρίσιμο όταν εξετάζουμε το θέμα της διεθνής μετανάστευσης και των διεθνών μεταναστών να μην κάνουμε να μην οδηγούμαστε σε αυτό το συμπέρασμα το οποίο είναι εντελώς σαθρό ότι εφόσον είμαστε γενναιόδοροι απέναντι στους παράδειγμους μετανάστες αυτό θα προσελκύσει και άλλους. Οποιοςδήποτε διαβάσει ε, κοινωνιολογικές μελέτες, ε, οικονομικές ε, σοβαρές μελέτες θα αντιληφθεί ότι η απόφαση που παίρνει κάποιος για να φύγει από τη χώρα του έχει να κάνει με προσωπικούς παράγοντες, προσωπικά στοιχεία και το τι τον περιμένει στη χώρα προορισμού δεν είναι βασικό κίνητρο. Μπορεί και να μην είναι καθόλου κίνητρο. Η απόφαση παίρνεται με την κατάσταση στη χώρα προέλευσης με βάση επίσης κάποιες πολιτιστικές, οικογενειακές, γλωσσικές συγγένειες. Αυτά έρχονται πολύ, πολύ πριν από το κίνητρο του πώς το μεταχειρίζεται κάποιος. Και κάτι ακόμα για αυτή την ιδέα για το ευρύτερο φάσμα. Όταν εξετάζουμε τα ζητήματα αυτά, είναι κρίσιμη σημασία να μην τα βλέπουμε όλα άσπρο-μαύρο. Είναι ευρύ το φάσμα σε επίπεδο λύσεων. Ο παράτυπος χαρακτήρας, παραδείγματο Χάριν μπορεί να αφορά κάποιον ο οποίος έρχεται σε μία χώρα παράνομα, με πλαστό διαβατήριο, ε, κρύβοντας την πραγματική ταυτότητα, ενώ πρόκειται για άτομα με κλιματικό παρελθόν, ε, και όπου η μόνη απάντηση είναι να σταλεί πίσω ο άνθρωπος τους, να πελαθεί για, για να μετομιστεί τέτοιου είδους παρατυπία ε, δεν μπορούμε να κάνουμε το ίδιο με κάποιον ο οποίος τέλειωσε η τουριστική του βίζα χθες και δεν έχει φύγει ακόμα από τη χώρα από ότι είναι παράτυπος εκείνη τη στιγμή. Στα Ηνωμένα Έθνη υπάρχουν σημαντικές μερίδες πληθυσμού, 11-12 εκατομμύρια άνθρωποι χωρίς χαρτιά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι οποίοι κατά τα λοιπά όμως επί δεκαετίες ε, είναι απόλυτα νομοταγείς. Εργάζονται, εκπαιδεύουν τα παιδιά τους, συμμετέχουν στο μέτρο του δυνατού στην ζωή της κοινότητάς τους. Έτσι λοιπόν εδώ είναι θέμα του ποια θα πρέπει να είναι η καταλληλότητα της απάντησης και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία αυτά. Οι απαντήσεις δεν πρέπει να ειδωθούν ως είτε θα του δώσουμε την ηθαγένεια είτε θα τον απελάσουμε. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες ε, έτσι ώστε να υπάρξει μια κάποια μορφή νομιμοποίησης. Να έχει κάποιος βασική πρόσβαση ε, στην εκπαίδευση, ε, στην περίθαλψη. Στις ομοσπονδιακές χώρες ε, ορισμένες φορές υπάρχουν και κάποια ε, στεγανά μεταξύ μετανάστευσης, αρχών μετανάστευσης, ε, αστυνομικών αρχών. Υπάρχουν, εν τόση, υπάρχει μια βεντάγια μέτρων, έτσι ώστε κάποιος κάποια στιγμή να φτάσει έως και την ηθαγένεια. Το χειρότερο πάντως πράγμα που θα μπορούσαμε να κάνουμε κατά το σχεδιασμό των πολιτικών αυτών είναι να εξετάσουμε μόνο αυτά τα δύο άκρα το, από την ηθαγένεια έως την απέλαση. Νομίζω πως θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα εάν μπούμε σε ένα δρόμο όπου σε 5 σε δέκα χρόνια θα μπορούμε να απαντούμε πιο κατάλληλα στην ιδιαιτερότητα του κάθε ανθρώπου, ε, της κάθε χώρας, χώρες οι οποίες κατά διαστήματα ήταν χώρες μετανάστευσης ε, και σε άλλα διαστήματα χώρες ε, προέλευσης, χώρες προορισμού. Θα αυξηθεί σημαντικά αυτό το φαινόμενο. Είναι η αρχή μιας διαδικασίας όπου τα πράγματα θα πάνε καλύτερα εάν όντως ακολουθήσουμε ένα δρόμο όπου θα μπορούμε να απαντούμε ε, πιο εμπεριστατωμένα απέναντι σε ένα περίπλοκο φαινόμενο. Αυτό θα ήταν επωφελές για όλους μας. Αυτά είμαι έτοιμη να απαντήσω στα ερωτήματά σας. Thank you, uh, for your... Ευχαριστώ κύριε Άρμπορ. Πολύ ενδιαφέρουσα η ομιλία σας. Έχουμε περίπου 45 λεπτά για τη συζήτηση ερωταπαντήσεις. Pardon? Okay. Um, so, please... Λοιπόν, παρακαλώ, ζητήστε το λόγο, αν θέλετε να μιλήσετε. Προς το παρόν έχουμε πέντε συναδέλφους εγγεγραμμένους. Θα προσπαθήσουμε να σημειώσουμε τα ονόματά σας. Θέλουμε να ακούσουμε όσο γίνεται περισσότερες απαντήσεις. Ε, θα περιορίσω το χρόνο αγόρευση, ένα δίλεπτο αν συμφωνείτε. ΕΛΚ, Κύριε Σχόλτη, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Τι να πω σε δύο λεπτά. Ευχαριστώ, κυρία Άρβορ, που ήρθατε. Εγώ είμαι από την Ουγγαρία, Ευρωβουλευτής και μέλος της Επιτροπής Ανάπτυξης, ΔΕΒΕ. Προσπαθώ λοιπόν να είμαι όσο γίνεται πιο κοντά στους ανθρώπους, επιτόπους, στις τοπικές κοινωνίες. Ας πούμε, έχουμε δώσει υποτροφίες σε 25 φοιτητές από περιοχές του Ιράκ και της Συρίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το στοιχείο της εκπαίδευσης. Θέλω όμως να σας κάνω τρία ερωτήματα συγκεκριμένα. Πρώτον, γνωρίζετε μια δήλωση 12 σημείων της χώρας μου η οποία έχει διανεμηθεί στη Νέα Υόρκη την περασμένη εβδομάδα. Αυτά τα 12 σημεία υπογραμμίζουν κάποια προβλήματα που υπάρχουν σε ευρωπαϊκές χώρες, σε ευρωπαϊκούς λαούς. Και θέλω να σας αφέρω δύο μόνο από αυτά. Πιστεύετε ότι το δικαίωμα στη μετανάστευση είναι θεμελιώδες δικαίωμα ή όχι. Για μένα είναι κρίσιμο ερώτημα αυτό. Δεύτερο ερώτημα. Τι πιστεύετε για το ρόλο του δικαιώματος στην παραμονή και του δικαιώματος στην επιστροφή. Διάβασα και τις 25 σελίδες πολύ προσεκτικά, αλλά είναι πραγματική πρόκληση αυτό με τρόπο έμεσο, έμεσο, όχι άμεσο. Εάν δεν προωθήσουμε το δικαίωμα στην παραμονή στη χώρα ε, για να αναπτύξει κάποιος τη χώρα του και να τη βοηθήσει, σημαίνει ότι του σωθούμε στη μετανάστευση. Και είναι πολύ εύκολο κάποιοι να το κάνουν αυτό. Αν μου επιτρέψει ο Πρόεδρος, θέλω να πω το εξής. Ευχαριστώ. Έχω πάει στο Ερμπίλ στο, πριν από δύο χρόνια. Δεν ήταν ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία φορά. Και εκεί καταλάβαμε ότι οι ποσοστώσεις στην Ευρώπη τι σημαίνουν. Για το Ερμπίλ, για τους πρόσφυγες, ήταν πράσινη κάρτα. Έτσι το ερμηνεύουν. Και είναι τελείω διαφορετική ερμηνεία που δίνουν στις ποσοστώσεις εκεί και εδώ. Και αν δεν υπάρξει αρκετή προσοχή, αν δεν προσέξετε πολύ γρήγορα, μπορεί αυτό να οδηγήσει σε παρερμηνίες και να θεωρηθεί πρόσκληση η ποσόστοση και θα πρέπει να καταργηθεί κατά την άποψή μου. Αυτά είχα να ρωτήσω. Και μια που είστε μόνο ομιλητή από πλευρά του ΕΛΚ, σα έδειξα τέτοια επίκαια. Ευχαριστώ πολύ για τη γενναιοδορία σα. Ορίστε, είναι, είναι η ουγγρική ανεκτικότητα αυτή. Ε, ε, η κυρία Γκόμες από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Um, thank you for coming. Σας ευχαριστώ που ήρθατε κυρία Άρβορ και ελπίζω να τα πείτε έξω από τα δόντια και στις κυβερνήσεις, όπως είπε και ο Γενικός Γραμματέας για τις ε, νομικές τους υποχρεώσεις, για να μην πω τις ηθικές υποχρεώσεις, θα πρέπει να απευθυνθείτε και στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, γιατί τίνουν να το λησμονούν. Ε, πολύ ενδιαφέρον αυτό το εγχείρημα το ΟΗΕ αλλά είναι κατάφορες οι αντιφάσεις. Και θέλω να σας ρωτήσω, δεν βλέπετε μεγάλη αντίφαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την τακτική και νόμιμη μετανάστευση σε αυτή τη διαδικασία του χαρτούμ και της βαλέτας που σημαίνει ότι δίνουμε χρήματα σε καταπιεστικές κυβερνήσεις για να είναι ακόμα πιο καταπιεστικές και να μην φεύγει ο κόσμος. Ο Σαλί Μαχμούτ που είναι στη φυλακή και πάλι γιατί ήρθε να κρούσει το γόδωνα του κινδύνου για την πατρίδα του, το Σουδάν και θα μπορούσα να φέρω και την Αιθιοπία και την Ερυθρέα κτλ. Τουρκία επίσης Πώς τη βλέπετε αυτή τη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία. Δεν είναι αυτό επαναπροώθηση, ρεφουλμό, κατά παραβίαση των υποχρεώσεών μας. Και μετά, η γαλάζια κάρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι ένας ασφαλής νόμιμος τρόπος μετανάστευσης. Αυτό είναι δουλειά για τους διακινητές, το είπε και ο Τόνιο Γκουτέρες. Αυτοί διαχειρίζονται αυτή τη στιγμή τις μεταναστευτικές ροές. Γιατί δεν υπάρχουν άλλοι νόμιμοι τρόποι να έρθει στην Ευρώπη από το να πέσει στα νύχια του διακινητή. Και τι πιστεύετε για αυτές τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις που δεν θέλουν να πάρουν μετανάστες και πρόσφυγες, αλλά πουλούν τα διαβατήριά τους με τις χρυσές θεωρήσεις διαβατηρίων και τα λοιπά σε πλήρη και κατάφορη και πάλι παραβίαση των κρατικών τους υποχρεώσεων αλλά και τις ευθύνες που έχουν να προστατεύουν τους πολίτες τους από την οργανωμένη εγκληματικότητα που τα εκμεταλλεύεται όλα αυτά. Φτωχούς μετανάστες δεν τους θέλουν, πλούσιους όμως τους πουλάνε και τις βίζες και τα διαβατήρια, δεν τους πειράζει. Ευχαριστώ. Η κυρία Βίξτρομ. start by wishing you... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχά να σα να σας καλωσορίσω θερμά στην, ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στη συνεδρίαση των επιτροπών μα. Ε, σα συγχαίρω για τη σκληρή δουλειά που εσεί και τα Ηνωμένα Έθνη γενικότερα κάνετε για την πολιτική μετανάστευση. Η μετανάστευση είναι πραγματικά όπω και εσεί τονίσατε ένα παγκόσμιο φαινόμενο και χρειάζεται να φέρουμε επιτάπητος παγκόσμιες λύσεις έτσι ώστε μιας και διαπαντός να επιλύσουμε όλα τα προβλήματα που σχετίζονται με τη μετανάστευση τόσο την νόμη μετανάστευση όσο και την μετανάστευση ασύλου. Για μένα προσωπικά ήταν μέγα προνόμιο να είμαι παρούσα στην διάσκεψη κορυφής όταν υπογράφηκε η δήλωση του ΟΗΕ και ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω πως όλοι χρειάζεται να ε, βασιστούμε σε αυτή την επιτυχία για να συνεχίσουμε. Βεβαίως ε, θα πρέπει να υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως μια στεναρή και ενωμένη φωνή και πάλι ε, με λύπησε που άκουσα ότι η Ουγγαρία, ένα κράτος μέλος, έχει πάλι δημιουργήσει δυσκολίες στη συζήτηση. Και πραγματικά ελπίζω πως θα μπορέσουμε να επανέλθουμε σε μια θέση όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να είναι ενωμένη και ισχυρή και να στηρίξει αυτό το, αυτή τη διαδικασία που τόσο πολύ χρειάζεται στον κόσμο. Βεβαίω, στην Ένωση θα πρέπει να μπορούμε επίση να συμβάλλουμε αναλαμβάνοντας το δίκαιο μας μερίδιο τη ε, της παγκόσμιας ευθύνης γιατί είμαστε σημαντικό κομμάτι του κόσμου και ως προς αυτό προσπαθείτε πολύ σκληρά αυτή τη στιγμή να επιφέρετε μεταρρυθμίσει για το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου. Εγώ είμαι εισηγήτρια για τη μεταρρύθμιση του κανονισμού του Δουβλίνου και είμαι εξαιρετικά περήφανη που τουλάχιστον εδώ μπορέσαμε χάρη σε μια εξαιρετική συνεργασία με τους συναδέλφους από πέντε από τις μεγαλύτερες ομάδες να καταφέρουμε ε, πλειοψηφία των δύο τρίτων του σώματος για μια πολύ φιλόδοξη μεταρρύθμιση. Είμαι πεπισμένη πως από κοινού θα αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και η κυρία Άρμπορ θα ήθελα να σας ε, διαβεβαιώσω ότι το Ευρωκοινοβούλιο και η Επιτροπή πάντοτε θα σας στηρίζει και θα συμμετέχει στη διαδικασία. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ κυρία Βίξτρομ. Τώρα εξ ονόματος των Πρασίνων η κυρία Λόχμπίλερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ ε, κυρία Λουίζα για την εξαιρετική σας δήλωση και σας ευχαριστώ που εξ αρχής τονίσατε σε αυτό το πολιτικό σώμα ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ενημέρωση βασισμένη σε στοιχεία ώστε να μπορούμε να χαράζουμε σωστά τις πολιτικές μας πράγματα το οποίο συχνά εμείς οι πολιτικοί το ξεχνάμε. Είπατε ότι Είπατε ότι το Παγκόσμιο Σύμφωνο είναι μόνο η αρχή. Πού βλέπετε να προχωράει η Σύμβαση της Γενέβης, γιατί στη χώρα μου κάποιοι λένε ότι η Σύμβαση της Γενέβης ίσως να είναι ξεπερασμένη. Επίσης, εδώ έχουμε και μια πτυχή ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εσείς είστε ειδικοί εμπειρογνώμονα σε αυτά τα θέματα. Πέρα από τα όσα ήδη μας είπατε, μπορείτε να ε, αναλύσετε περισσότερο ε, Πού βλέπετε να βρίσκονται τα ανθρώπινα δικαιώματα σε αυτή τη διαδικασία. Και επίση θα ήθελα να γνωρίζω ποια είναι η κρίση σα για την Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία, ειδικά με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τελευταία μου ερώτηση. Είπατε ότι είστε στην διαδικασία της διαβούλευσης. Φαντάζομαι ότι ΜΚΟ και οι βουλευτές είναι ευπρόσδεκτοι να συμβάλλουν. Όμως στην ίδια τη συνεδρίαση στο Μαρακές υπάρχει ένα είδος φόρουμ των ΜΚΟ ή άλλες δυνατότητες πέρα από τις επίσημες συνεδριάσεις ώστε να μπορεί κανείς να συμβάλλει στη συζήτηση. Ευχαριστώ Μπάρμπαρα Λοχμπίλερ και για να κλείσουμε τον πρώτο γύρο παρεμβάσεων θα δώσω το λόγο στον κύριο Πετίδιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να καλωσορίσω και εγώ την κυρία Άρμπουρ και να τη θέσω κάποιε ερωτήσει, επειδή δεν αναφέρθηκε στα συγκεκριμένα θέματα κατά τη διάρκεια τη ε, ενημερώσεώ τη. Θα πρέπει, προκειμένου να γίνουν αποδεκτοί κάποιοι μετανάστες, τα κράτη να λαμβάνουν υπόψη το κριτήριο της δυνατότητας να απορροφήσουν συγκεκριμένο αριθμό μεταναστών και αν αυτό το όριο έχει ξεπεραστεί όπως συμβαίνει στην πατρίδα μου την Ελλάδα, τι πρέπει να γίνει εκεί. Θα πρέπει να εξακολουθούν να έρχονται και άλλοι μετανάστες ή πρέπει να τους στείλουμε σε κάποια άλλη περιοχή που μπορεί να τους απορροφήσει. Ένα δεύτερο ερώτημα είναι αν τα κράτη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη προκειμένου να αποδεχτούν κάποιο μετανάστη την διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στη θρησκεία και στην ε, πολιτισμική κληρονομία των ανθρώπων αυτών με τους γηγενείς. Ένα τρίτο ερώτημα είναι εάν θα πρέπει ένα κράτος να έχει τη δυνατότητα να αρνείται να δεχθεί κάποιους μετανάστες εάν πιστεύει ότι η είσοδός θα δημιουργήσει προβλήματα ασφαλείας και αυξήσεως της εγκληματικότητας στη χώρα της υποδοχής. Και τέλος, ποια είναι η θέση σας απέναντι στην τακτική της Τουρκίας να προωθεί κατά χιλιάδες παράνομους τους μετανάστες προς την Ευρώπη μέσω της Ελλάδος. Ευχαριστώ. Thank ε, Ευχαριστώ. Κυρία Άρμπορ, θα θέλετε να απαντήσετε σε ένα πρώτο γύρο, να συνεχίσουμε με δεύτερο γύρο, τι προτιμάτε. Ίσως να απαντήσω τώρα σε αυτό το πρώτο γύρο. Παρακαλώ. Έχουμε πολλούς ακόμα συναδέλφους που αγωνιούν να κάνουν ερωτήσεις. είμαι πάρα πολύ σύντομη. Για την πρώτη ερώτηση. Γνωρίζω τα 12 σημεία που επέβαλε, ε, υπέβαλε συγγνώμη, η Ουγγρική κυβέρνηση. Στο δεύτερο γύρο θα συζητηθούν. Ε, ο Υπουργό Εξωτερικών. Έχω κάποια ανησυχία. Τα 12 σημεία φαίνεται να ε, σηματοδοτούν μια θέση ε, των Ηνωμένων Εθνών. Μα δεν υπάρχει ακόμα ενιαία θέση των Ηνωμένων Εθνών για τη μετανάστευση. Πολλές είναι και υπηρεσίε σε οργανισμοί 22 των Ηνωμένων Εθνών, συν ε, το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, που ασχολούνται με θέματα μετανάστευσης και όλα αυτά τα χρόνια έχουν κατευθυντήριες γραμμές, διαδικασίες, ε, πρότυπα κτλ. Ο Γενικός Γραμματέας εξέδωσε τη δική του έκθεση αρχές Ιανουαρίου, που προβάλλει τη δική του άποψη και το δικό του όραμα για τη μελλοντική μεταχείριση της μετανάστευσης και το Παγκόσμιο Σύμφωνο που διαπραγματευόμαστε είναι η ιδιοκτησία των κρατών μελών και θα αποκτήσει τη μορφή που θα θελήσουν να του δώσουν τα κράτη. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει προώθηση της μετανάστευσης από το Ηνωμένα Έθνη ούτε κανένα ενιαίο έγγραφο. Διαπραγμάτευση γίνεται για το Παγκόσμιο Σύμφωνο. Ο Γενικός Γραμματέας όντως έχει κάνει κάποιες προτάσεις προσωπικές. Τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ είναι εκείνα που θα αποφασίσουν αν θα το προωθήσουν αυτό το θέμα. διστάζω πάρα πολύ ε, να εκφράσω νομικές απόψεις. Ήμουν ε, δικαστή στο Νότο Δικαστήριο του Καναδά. Όταν εκφράζει κάποιες νομικές απόψεις θα πρέπει να είναι συγκρατημένος και προσεκτικός, αλλά στο Διεθνές Δίκαιο και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ο καθένας έχει το δικαίωμα να φύγει, να παραμείνει, ή να διαπανέλθει στη χώρα του. Αυτό είναι μια βασική αρχή και ένα πλαίσιο που διέπει την κινητικότητα. Τώρα τι σημαίνει έχεις το δικαίωμα να φύγεις από μια χώρα όταν δεν έχεις δικαίωμα να μεταβείς κάπου αλλού, τι σημαίνει αυτό. Θα μπορούσαμε τώρα να κάνουμε διάφορες εικασίες για το φάσμα που καλύπτει αυτό το ε, δικαίωμα, αλλά δεν θέλω να εκφέρω νομική άποψη. Στην έκθεση του Γενικού Γραμματέα, τι αναφέρεται, υπερασπίζεται πάρα πολύ ε, τη διάνοιξη περισσότερων νομίμων οδών όχι ως μόνο τρόπο, αλλά ως ένα ευφυή τρόπο να ε, παταχθεί η παράτυπη μετανάστευση και να παρακαυθεί. Σε κάποιες ερωτήσεις που έγιναν ε, αναφέρθηκαν ε, οι μετανάστες και οι πρόσφυγες συγκεκριμένα κάπως. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι σε ένα περιβάλλον όπου είναι πάρα πολύ λίγες οι νόμιμες οδοί, οι περισσότεροι που χτυπούν την πόρτα σας θα ζητήσουν άσυλο. Γιατί είναι ο μόνος τρόπος να βρεθεί νόμιμος τρόπος για να μπουν στη χώρα. Αυτό το είδαμε στην κρίση που γνώρισε η Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Πάρα πολλοί ε, άνθρωποι, πάρα πολύ συχνά ε, και μικτές, μικτά κύματα προσφύγων και μεταναστών φτάνουν στις πόρτες της Ευρώπης. Και επειδή ε, τότε ο μοναδικός τρόπος ήταν το άσυλο, ο μόνος τρόπος να ζητήσουν νόμιμη είσοδο, ζητούσαν άσυλο. Το πρόβλημα είναι ότι απορρίπτονται ε, αυτές οι αιτήσει γιατί ε, δικαιούνται μόνο οι πρόσφυγες με βάση τη Σύμβαση Γενέβης του 1951. Ε, όσοι προσπαθούν να ξεφύγουν από τη δίωξη. Αλλά τώρα ο κόσμος ξεφεύγει από τον πόλεμο, δεν ε, είναι προσωπική ε, δίωξη κάποιο από μια κρατική αρχή, αρχή ασφαλείας ε, Σύρια ας πούμε και κάποιοι που έρχονται από άλλες ε, χώρες κατάφεραν να πάρουν πιο συχνά άσυλο από ό,τι άλλους και ορισμένοι δεν μπόρεσαν να αποδείξουν ότι διώκονται. Γι' αυτό υπήρχαν πολλές και πολλά προβλήματα επιστροφών για τα ευρωπαϊκά κράτη. Για ορισμένοι, για από εκείνους, δόθηκε ε, προσωρινή άδεια παραμονή σε χώρες που επιθυμούσαν να παραμείνουν για να ανοίξουν περισσότερες νόμιμες οδοί για την κανονική μετανάστευση, την συντεταγμένη κτλ. Για να παραμένουν στη χώρα με τρόπο συντεταγμένο και νόμιμο, που εργάζονται στην κανονική πραγματική οικονομία και όχι στην παραοικονομία, όπω συμβαίνει συχνά. Εργάζονται βεβαίω. σε άλλε περιπτώσει, στην παραοικονομία ή στη, μαύρη αγορά όπως αναφέρει. Αυτό δεν είναι λύση που να επέβαλε κανείς σε κανέναν. Η διαδικασία του ΟΗΕ είτε είναι η έκθεση του Γενικού Γραμματέα είτε το σύμφωνο που διαπραγματευόμαστε σε καμία περίπτωση ε, δεν έχει στόχο να επιβάλλει οποιοδήποτε μοντέλο σε κανένα. Είναι ε, μια διαπραγμάτευση προς ένα έγγραφο σύμφωνο που δεν είναι νομικά δεσμευτικό, που θα παρέχει μια σειρά επιλογών αλλά ε, ελπίζουμε ότι θα ανοίξει την πόρτα για διάφορους τρόπους να υποστηρίξουμε την ασφαλή και συντεταγμένη και νόμιμη μετανάστευση, αποθαρρύνοντας και αποτρέποντας την ε, επικίνδυνη παράτυπη μετανάστευση. Θα ήθελα να τονίσω ότι έχουν γίνει πάρα πολλές συζητήσεις, γιατί με ρώτησε κάποιος για τη Σύμβαση Γενέβης, αν θα πρέπει να ξανανοίξουν όλες για το δίκαιο του πολέμου ή μόνο για τους πρόσφυγες. Για τη μετανάστευση θέλω να πω ότι στην αρχή της διαδικασίας αυτής ζητήθηκε να αναγνωριστεί ξεχωριστή κατηγορία κλιματικών μεταναστών που να τους χαρακτηρίζουμε πρόσφυγες. Αυτό ε, γνώρισε, μάλλον γέννησε μεγάλη συμπάθεια στην κοινή γνώμη, ιδιαίτερα όταν κατανοεί ο κόσμος ότι στην Ασία και στον ε, Ειρηνικό ε, ε, οι μικρές νησιωτικές χώρες είναι εκτεθειμένες και πραγματικά κινδυνεύει να πλημμυρίσει η χώρα και να χαθεί. Υπάρχει μια γενική λοιπόν συμπάθεια στα μάτια του κόσμου λόγω των φυσικών καταστροφών, θεομηνιών, από τσουνάμι, σεισμούς, γειτονικές χώρες που βοηθούν προσωρινά αυτό σίγουρα προφανώς θα πρέπει να εθαρρυνθεί. Αυτή τη στιγμή δεν είναι ξεκάθαρο εάν ε, μπορεί, αν θα πρέπει να ε, γίνει πιο επίσημο αυτό. Θα πρέπει να, να δούμε περισσότερο ε, την αναγκαστική εκτόπιση. Τι είναι η αναγκαστική μετανάστευση, πώς ορίζεται η εθελούσια, η, η εκούσια, η ακούσια, τι γίνεται με την κλιματική αλλαγή, την απερίμωση, πότε θεωρείται η μετανάστευση ως αναγκαστική και όχι ως προαιρετική ή ακούσια. Όλα αυτά αυτή τη στιγμή δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστούν στο παρόν εγχείρημα. Γι' αυτό λέω ότι τώρα βρισκόμαστε μόνο στην αρχή μια διαδικασία. Όπως το 1992 που ήταν παγκόσμια Σύνοδο κορυφής για τη γη, για τον πλανήτη, ε, αφύπνισε τις συνειδήσεις ε, σχετικά με το περιβάλλον και μετά ε, από 20 χρόνια και πλέον φτάσαμε στη Συμφωνία του Παρισιού. Βρισκόμαστε λοιπόν σε ένα πάρα πολύ πρώιμο στάδιο στην παρούσα διαδικασία. Υπάρχει μεγάλος χώρος για τον ιδιωτικό τομέα, την κοινωνία των πολιτών, τους βουλευτές. για να συμμετέχουν ε, όσοι δεν είναι εκπρόσωποι κυβερνήσεων. Σε κάθε γύρο διαπραγματεύσεων στη Νέα Υόρκη υπάρχει χρόνος που έχει προβλεφθεί για τη συμμετοχή ε, διαφόρων ενεχομένων πολλαπλών που δεν είναι κυβερνητικοί και φυσικά θα δοθεί ε, στη διάσκεψη του Μαρόκου άπλετος χώρος και χρόνος αυτούς όταν θα εγκριθεί το Παγκόσμιο Σύμφωνο μετά τη λήξη των διαπραγματεύσεων τον Ιούλιο. Δεν μπορώ παρά να επαναλάβω και πάλι ότι αυτό το παγκόσμιο σύμφωνο δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση επιβολή οποιασδήποτε ειδική μεταναστευτική πολιτική σε μια χώρα με στόχου, αριθμού, ποσοστώσει. Απευθύνεται σε ολόκληρο τον κόσμο και σε μέρη του κόσμου, ας πούμε στις χώρες του κόρπου, όπου 80% ε, του πληθυσμού είναι ξένοι εργάτες, ε, όπως άλλες χώρες, ας πούμε, στις Φιλιππίνες, στο Μπαγκλαντές, που έχουν πάρα πολύ ε, μεγάλες κοινότητες μεταναστών εργαζομένων που εργάζονται στο εξωτερικό και περιμένουν να τους βοηθήσουν να επιστρέψουν στις χώρες τους κάποια στιγμή μετά από 5, 10, 15 χρόνια. Ε, αυτά τα θέματα έχουν διάφορες όψεις και μορφές. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι που έχει να κάνει με τη διαπραγμάτευση της Σύμβασης της Γενέβης. Υπάρχει ένα καθεστώς διεθνούς προστασίας που θα πρέπει όλοι να επεκτείνουν όλα τα κράτη-μέλη σε εκείνου που είναι πρόσφυγες, που είναι γύρω στα 25 εκατομμύρια και δικαιούνται να ζητήσουν άσυλο και δικαιούνται διεθνούς προστασίας. Ευχαριστώ. Έχουμε χρόνο για ένα δεύτερο γύρο τώρα. We go down to one ένα λεπτό όμω, Τώρα υπάρχει περιπτώσει όσο γίνεται πιο σύντομη. Να είστε κυρία Γερόκα από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ για τι απαντήσει και για την παρουσίασή σα. Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποιε μελέτε που έχω κάνει ω ανθρωπολόγο. Ασχολούμαι με, με, με τις κοινότητες του 1992, από τότε που έφτασαν οι πρώτοι Ρωμά στην Γερμανία. Ήταν η Γερμανία η μόνη χώρα που υποδεχόταν τότε τους βαλκανικού πολέμου και μάθαμε ε, και με τους ε, Τούρκους ε, στη Γερμανία, ε, ποια είναι, ποιος είναι ο τρόπος της ένταξης και για τους Ρωμά. Και είχαμε βεβαίως και άλλους μετανάστες έκτοτε. Θα ήθελα να ρωτήσω ποια είναι τα δικά σας ευρήματα διότι τα τελευταία δύο χρόνια στα διάφορα, στους καταβλισμούς στην ε, ε, Γερμανία, στη Γαλλία, στην Αγγλία, στην Αυστρία, στην Ελλάδα έχω πάει εγώ, έχω πάει στους, στα στρατόπεδα τα, τα μεταναστευτικά και αυτό που βλέπουμε είναι ε, ότι όχι μόνο οι μετανάστες τρίτης γενιάς, οι φίλοι μου που τους ξέρω από μικροί, αλλά και άλλοι που είναι εδώ και περιμένουν μια απόφαση τους στέλνουν με τους όρους στην Εσθονία παραδείγματος χάρη γυρίζουν πίσω κρυφά στη Γερμανία ε, τα παιδιά τους δεν τους δίνουν να φάνε στα σχολεία εκεί ε, ποιες είναι οι απαντήσεις μας λοιπόν απέναντι στις, κοινότητες ε, ε, που υποδέχονται τους ανθρώπους αυτούς. Ε, οι παιδαγωγικές, οι κοινωνιολογικές ε, απαντήσεις. Στην Ουγγαρία ως κι, κοινωνιολόγος έχω επισκεφθεί κέντρα μεταναστών. Έχουμε δει την ένταξη των ανθρώπων που όταν πάνε κάπου εκεί που θέλουν να πάνε στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για του Ρωμά, παραδείγματο χάρη, είχαμε επικεντρωθεί σε αυτέ τι ομάδε των 5 εκατομμυρίων ανθρώπων περίπου. Ε, Πώ βλέπετε το μέλλον, Διότι μόνο έτσι θα μπορούσαμε, θα μπορούσαμε να δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια για του υπόλοιπου που θέλουν να έρθουν. Ευχαριστώ. Η κυρία Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ την Λίζα Άρμπορ για την παρουσία της σήμερα εδώ. Είναι πολύ σημαντικό και το γεγονός ότι επανέλαβε το γεγονός ότι αυτό το έγγραφο θα πρέπει να εστιάσει περισσότερο στους ανθρώπους. Ε, ακριβώς ε, βλέπουμε πόσο πολυδιάστατο είναι αυτό το φαινόμενο τη σημασία της συνεργασίας, δηλαδή ευθύνη των κρατών μελών, όπως το επανέλαβαν και άλλοι συνάδελφοι. Τα κράτη-μέλη οφείλουν να μοιραστούν στις ευθύνες τους για να μπορέσουν να διαχειριστούν το φαινόμενο μέσα από την ελληνική. Η Ατζέντα 2030 για την, για την βιώσιμη ανάπτυξη και να περάσω σε άλλο σημείο ότι το έγγραφο αυτό είναι ένα πλαίσιο μη δεσμευτικό για συνεργασία. Γι' αυτό τον λόγο οι αρχές, οι κατευθυντήριες ε, θα πρέπει να μείνουν απαράλλακτες στη διάρκεια της φάσης της διαπραγμάτευσης. Αναφέρομαι ιδιαίτερως στο κεντρικό ρόλο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την ασφάλεια, της ασφάλειας, την αξιοπρέπεια των μεταναστών και των προσφύγων. Να τονίσουμε επίσης στην αρχή της μη, της μη ε, του non-refoulement ε, και να κλείσω ζητώντας ένα σχόλιο από πλευρά σας, ε, κυρία Άρμπορ, για τα όσα συνέβουν. Ας πούμε, το ισπανικό πλοίο που έσωσε 250 μετανάστευσες και ε, κατηγορείται για συνεργασία σε αδίκημα, ακριβώς επειδή ε, βοήθησε ανθρώπους να μην πνιγούν. Λάμπερτ. Ευχαριστώ πολύ για την εισήγησή σας και για τα όσα μόλις λέγατε για τους κλιματικούς πρόσφυγες και τους εκτοπισμένους λόγω κλιματικών αλλαγών. Εγώ θέλω να αναφερθώ σε ένα άλλο σημείο που είπατε κι εσείς σε σχέση με το πώς θα μπορούσαμε να έχουμε θετικές εμπειρίες για περισσότερο κόσμο. Άρα, τι έμφαση πιστεύετε ότι θα πρέπει να δοθεί Ας πούμε, στην πρόσφατη ατζέντα του Παγκόσμιου Οργανισμού Εργασίας ή ε, τη σύμβαση του ΑΕΛΟ για τους οικιακούς εργαζόμενους. Έπειτα, για τα όσα λέγατε, εγώ λίγο αλλάζω την ε, διαπίστωση η Ευρώπη θα πρέπει να καταλάβει ότι δεν έρχονται και όλοι στην Ευρώπη και ότι η μετανάστευση νότου-νότου είναι εξαιρετικά σημαντική επίσης. Τι θα μπορούσαμε να πούμε για ε, τις περιφερειακές συμφωνίες όπως για παράδειγμα τις ρυθμίσεις που έχει κάνει η Σρι Λάγκα ώστε να σταματήσει τις γυναίκες που εργάζονταν ως οικιακές βοηθείς στη Σαουδική Αραβία εκτός αν άλλαζαν οι συνθήκες εργασίας τους ή αυτό που λέμε εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο τους ε, ε, Μπαγκλαντεσιανούς που πάνε στο Κατάρ για να δουλέψουν, να χτίσουν τα στάδια για το παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Τι μπορούμε να κάνουμε δηλαδή ώστε η μετανάστευση να είναι πιο θετική εμπειρία για εκείνους που, είναι, που εργάζονται σε άλλες χώρες και να εστιαστούμε σε αυτό. Και όχι τόσο όπως κάνουμε εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, παράνομη και όχι παράτυπη ε, πτυχή όλου αυτού του φαινομένου. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα, αυτό που έχουμε είναι ένας κατάλογος από συναδέλφους σοσιαλιστών. Πέντε τον αριθμό. Ναι, είναι η πιο πολύ ομάδα εδώ. Ένα λεπτό ο καθένας, οπότε να οικονομήσουμε χρόνο και να έχουμε περισσότερο χρόνο για την απάντηση. Κύριος Κιώσλερ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Άρμπα. Και για τον υφάλαιο ε, τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται τα πράγματα αντικειμενικά και πραγματικά πολύ ευεργετικά. Να ε, δούμε λίγο την κατάσταση στη Λιβύη, γιατί έχουμε ειδική σχέση με την κατάσταση αυτή. Μέχρι τώρα υπάρχει μια εκθέση που δεν έχει δημοσιευτεί των Ηνωμένων Εθνών όπου ε, γίνεται λόγος για βασανιστήρια ε, από πλευράς ε, των δυνάμεων ασφαλείας της ενίας κυβέρνησης της Λιβύης. Αυτή η αδημοσίευτη έκθεση λοιπόν κάνει λόγο για βασανιστήρια, για δουλεμπόριο, αυθαίρετες συλλήψεις και προσφύγων και βεβαίως όλα αυτά διαπράττονται από μια επίλεκτη ε, μονάδα σώμα ε, της Λιβικής κυβέρνησης που υπάγεται άμεσα στο Υπουργείο Εσωτερικών. Γίνεται λόγος και ε, από μία ψυχολόγο που κοιτάει αυτούς τους πρόσφυγες και λέει ότι μαθαίνουμε ότι στα κάμπ της Λιβύης υφίστανται ξυλοδαρμούς, βιασμούς, από τους διακηρυτές, παίρνουν τους γονείς του τηλέφωνο με ένα μαχαίρι στο λαιμό λέγοντας αν δεν στείλει αμέσως λεφτά θα το σφάξω ή θα τη σφάξω ε, την κόρη σου και το γιο σου. Και πάρα πολύ ε, σεξουαλική βία, ε, ξυλοδαρμή, ε, και καίνε με τσιγάρα διάφορα φρικτά πράγματα. Πότε θα δημοσιευτεί αυτή η έκθεση για να συζητηθεί αντίστοιχα επίσημα και στο Κοινοβούλιο και να λάβουν γνώση οι βουλευτές. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φρόιντ. Πού είναι το μικρόφωνο. Εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς θα ήθελα να σας πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω πέντε γυναίκες να κάθονται εκεί στο πάνελ που δεν είναι καθημερινό φαινόμενο στο κοινοβούλιο. Ορίστε, μας βγήκε και φεμινιστής. Ε, ε, και... Ε, έχουμε και, τον πρόεδρο βέβαια. Ε, δεν είναι πρόβλημα των σοσιαλιστών, κύριε Πρόεδρε, ότι είναι πέντε παρόντες και ζητούν το λόγο. Είναι το πρόβλημα του ΕΛΚ που απουσιάζει και δεν ενδιαφέρεται μάλλον για το θέμα. Δεν φταίμε εμεί που είμαστε παρόντες και ενδιαφερόμαστε. Λοιπόν, τι έλεγα. Η ερώτησή μου έχει να κάνει με αυτό που είπατε εσείς κύριε Άρμπορ και πραγματικά το εκτίμησα πάρα πολύ ε, όλη την ομιλία σας. Λέτε ότι ξεκινάμε από λάθος συμπέρασμα ε, ότι αν είμαστε γενναιόδοροι ε, και σωστοί στη συμπεριφορά μας θα έρθουν περισσότεροι παράτυποι μετανάστες. Όπως γνωρίζετε σε όλες τις χώρες που έχουν δεχτεί πολλούς μετανάστες κυριαρχεί αυτό το επιχείρημα. Ακόμα και χώρες που δεν πήραν κανέναν μετανάστη είπαν «Ε, μόλις υποδεχτούμε κάποιους θα έρθουν και όλοι οι υπόλοιποι. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, Θέλετε να επεκταθείτε λίγο παραπάνω. Ε, πώς καταρρύπτεται αυτό το επιχείρημα. Αναφερθήκατε επιγραμματικά σε αυτό. Θα ήθελα λίγο περισσότερο να μας πείτε. Ευχαριστώ πολύ. Η Τάνια Φαγιόν. Thank you. Chair and... Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να σα ευχαριστήσω για τις εισφορέ σα, τα σχόλιά σα για το να ότι είστε εδώ μαζί μα σήμερα. Έχω δύο ερωτήματα. Νομίζω ότι δεν αναφερθήκατε σχετικά έως τώρα. Ε, θα ήθελα να ξέρω πώς εκτιμάτε εσείς την απόσυρση της Αμερικανικής κυβέρνησης από τις διπραγματεύσεις ε, για το Παγκόσμιο Σύμφωνο. Πιστεύετε ότι θα υπάρξουν επιπτώσεις θα υπάρξει αντίκτυπος και κάτι άλλο που είναι εξαιρετικά σημαντικό. Το θέμα των περιβαλλοντικών μεταναστών, των προσφύγων για κλιματικούς λόγους, είναι μια έννοια την οποία ακόμα ε, δεν έχουμε καταφέρει ε, να προσδιορίσουμε, δεν έχουμε μπορέσει να τους περιλάβουμε σε κείμενα. Εσείς πώς ε, πιστεύετε ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό, το πολύ σημαντικό θέμα για το μέλλον. Ευχαριστώ, Τάνια Ανελίτς. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Και πέρσι δοθήκαμε στη Νέα Υόρκη με τη Λίντα Μακάβαν με θέμα του στόχου τη ε, χιλιετία, ε, τη βιώσιμη ανάπτυξη μάλλον και του πρόσφυγε. Θέλω να ρωτήσω και εγώ για του κλιματικού πρόσφυγε, γιατί αυτό τον καιρό εκπονώ μια έκθεση ε, για την διπλωματία του κλίματο ε, και έγινε μια συζήτηση με τους σκιώδεις ηγητές όπου δεν θεωρήθηκε σκόπιμο να συμπεριληφθεί αυτός ο όρος. Καλύπτεται από το Παγκόσμιο Σύμφωνο, θα καλυφθεί η κατηγορία αυτή των κλιματικών προσφύγων. Γιατί δεν αναφέρεται πουθενά ακόμα ο όρος του κλιματικού πρόσφυγα. Ε, ε αναπτύσσεται κάποια δυναμική. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να προχωρήσουμε σε ένα ορισμό του τι εστί κλιματικός ε, πρόσφυγες και θα είναι δύσκολο να μπει και στη δική μου έκθεση για την κλιματική διπλωματία, αλλά θα με ενδιαφέρει η διαπάντησή σας. Ευχαριστώ, Αναλίτς. Τελευταία ομιλήτρια είναι η κυρία Σλάιν. Um, Ευχαριστώ. Είναι σημαντικό να γίνεται αυτή η συζήτηση με τη συμμετοχή των τριών αυτών επιτροπών. Πρέπει να εργαστούμε με πιο συντονισμένο τρόπο. Ανησυχώ κάπως ε, για το πώς αναπτύσσεται η πτυχή της μετανάστευσης. Πάμε όλο και πιο πολύ προς, τα, ζητήματα ασφάλειας ε, και ίσως ό,τι αφορά τη βοήθεια, την ενίσχυση, ε, τίθενται κάποια κριτήρια ασφαλείας ε, και αυτό δημιουργεί προβλήματα σε σχέση με τους στόχους ε, εκρίζωσης ε, των, ε, της φτώχειας. Ήμουν στη Συνόδο Κορυφή στην Αφρική με κάποιους συναδέλφους και το επίπεδο φιλοδοξίας ήταν υψηλό αλλά ελπίζω ότι το έργο σας θα βοηθήσει για να μειωθεί η υποκρισία που υπάρχει. Άλλα ακούμε στη Νέα Υόρκη και άλλα γίνονται σε εθνικό επίπεδο. Είναι σημαντικό να θυμίσουμε ότι αυτή η πρόκληση να, μοιραστούμε, να μοιραστούμε καλύτερα τις ευθύνε μας ε, σε ό,τι αφορά τους πρόσφυγες δεν αφορά μόνο την Ευρώπη, αφορά ε, τον κόσμο ολόκληρο. μπορούμε στο Παγκόσμιο Σύμφωνο ε, να πούμε κάτι ε, που να ε, μας βοηθήσει να αποφύγουμε την ποινικοποίηση των κυβερνικών οργανώσεων, διότι έχουμε πολύ αρνητικές εξελίξεις στο τελευταίο διάστημα προς την κατεύθυνση αυτή. Πρέπει να πούμε κάτι στο Παγκόσμιο Σύμφωνο για την ανάγκη να μην ποινικοποιούνται αυτοί που βοηθούν και να, δοθ, να δοθούν περισσότερα επίση και για την εταιρική σχέση την παγκόσμια για τι δεξιότητε. Ε, ευχαριστώ. Ε, δεν φαίνεται να θέλει κάποιο άλλος το λόγο. Ε, η κυρία Άρμπουρ για δεύτερη φορά, για δεύτερο γύρο απαντήσεων. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα απευθυνθώ στα ζητήματα αυτά έτσι κάπως πιο συμπυκνωμένα. ορισμένα είναι επιμέρους θέματα βέβαια και δεν μπορώ να πω κάτι ιδιαίτερο εγώ έγινε αναφορά στο θέμα της ένταξης των μεταναστών ε, στις ε, χώρες υποδοχής. Είναι μια πτυχή την οποία ε, αναφέρουμε στην έκθεση του, του Γενικού Γραμματέα. Θέλουμε ιδίως να εξασφαλίσουμε ότι όταν μιλάμε για βοήθεια στη μεταναστευτική διαδικασία πρέπει να δίνουμε μεγάλη έμφαση στις ανάγκες των κοινοτήτων υποδοχής. Οι πολιτικές μετανάστες συνήθως ε, αποφασίζονται σε εθνικό επίπεδο, αλλά σε τοπικό επίπεδο ζούμε τα αποτελέσματα της πολιτικής αυτής, της πόλης, στην περιφέρεια, της γειτονιές, όταν μετανάστες είτε είναι παράτυποι αλλά και νόμιμοι φτάνουν σε μια κοινότητα, ε, εγκαθίστανται συνήθως ε, στις πιο φτωχές περιοχές της χώρας υποδοχής. Είναι κρίσιμο, είναι σημαντικό, εάν θέλουμε να δημιουργήσουμε αρμονία ε, και όχι επιφυλακτικότητα και αρνητικά συναισθήματα μεταξύ των νεοαφιχθέντων και των κινητών υποδοχής, να ληφθούν υπόψη και οι ανάγκες των κοινοτήτων αυτών. Υπάρχουν πολλές πολιτικές ένταξεις που θα μπορούσαν ε, να ε, προωθήσουν μία στάση πιο θετική. Ε, βεβαίως οι ίδιοι αυτοί οι μετανάστες ε, μπορεί να αξίζουν καλύτερες μεταχείρισης, μπορεί να έρχονται από δύσκολες καταστάσεις, αλλά δεν θα βρουν αυτή τη μεταχείριση σε κοινότητες όπου ήδη υπάρχουν σημαντικά προβλήματα. Απέναντι λοιπόν και στους πρόφυγες και στους οικονομικούς μετανάστες, είτε είναι νόμιμοι είτε παράτυποι, το ίδιο ισχύει. Να πω κάτι και για την, το Διεθνή Οργάνωση Εργασίας ε, και τα, την αξιοπρεπή εργασία. Όταν μιλάμε για πενάστευση αμέσως, ε, αμέσως περνάμε στα αρνητικά, στο παθολογικό κομμάτι. Αυτοί οι 258 εκατομμύρια μετανάστες στον κόσμο, οι περισσότεροι από αυτούς έχουν ακολουθήσει ε, ασφαλείς διάβλους, νόμιμους διάβλους. Όμως, σε γενικές γραμμές αντιμετωπίζουν πολλών λογιών εμπόδια έχουν να κάνουν με τις, ε, ε τις εργασίες, τις ξενοφοβικές ε, στάσεις, ε, οι οποίες πυροδοτούνται ακριβώς από αυτήν την στάση απέναντι στους παράτυπους μετανάστες και όλοι επηρεάζονται από αυτές. Το θέμα των προτύπων λοιπόν της Διεθνής Οργάνωσης Εργασίας για την αξιοπρεπή εργασία, το θέμα του ενιαίου εργοδότη είναι ένα κρίσιμο ζήτημα, ε, ιδιαίτερα στις χώρες του κόλπου, όπου συνήθως ε, είναι συνδεδεμένος ο μετανάστης με έναν μόνο εργοδότη, ε, ο οποίος έχει τεράστια εξουσία επί του ανθρώπου αυτού. Η παρουσία εκεί εξαρτάται από αυτό. Προσπαθούμε αυτό το μοντέλο να το περιορίσουμε, ιδιαίτερα όταν είναι το μόνο μοντέλο σε μια χώρα. Ε, το θέμα επίσης των εργαζομένων ε, στα οικιακά, είτε είναι παράνομη, είτε, είτε είναι παράτυπη την νόμιμη μετανάστευση και στην περίπτωση αυτή, το θέμα αυτό πρέπει να καλύπτεται ε, στο Παγκόσμιο Σύμφωνο, τα άτομα δηλαδή τα οποία πολύ εύκολα μπορούν να γίνουν αντικείμενο καταχρήσεων. Ε, το θέμα των περιορισμών και των δικαιωμάτων των γυναικών να μεταναστεύσουν για λόγους εργασίας είναι ένα πολύ δύσκολο ζήτημα. Αφενός, όπως είπα νωρίτερα, ο κάθε πολίτης θεωρητικά έχει το δικαίωμα να παραμείνει, να εισέλθει ή να φύγει από μία χώρα. Το να παρεμποδίζουμε λοιπόν ε, τις γυναίκες εργαζόμενους που θέλουν να πάνε αλλού είναι παραβίαση του δικαιώματος αυτού. Ταυτόχρονα βεβαίως υπάρχει το ευάλωτος χαρακτήρας των νέων γυναικών που εργάζονται στον τομέα της περίθαλψης, ε, σε οικιακές εργασίες. Ε, είναι τεράστιες οι δυνατότητες ε, εκμετάλλευσης και γι' αυτό πολλές χώρες βάζουν κάποιο όριο ηλικίας ή κάποιους άλλους περιορισμούς. Δεν μπορώ να πω κάτι ιδιαίτερο τώρα για τη Λιβύη και τον παρόν διακανονισμό με τα Ηνωμένα Έθνη, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώς ε, δεν έχω επαρκή στοιχεία για να πω οτιδήποτε γι' αυτό. Πρέπει πάντως πάντα να θυμόμαστε ότι παρότι βεβαίως δίνεται μεγάλη έμφαση στο τι συμβαίνει στη Λιβύη, ε, υπάρχει και οργανωμένη βία και αλλού στον κόσμο, στην Κεντρική Αμερική, παραδείγματος χάρη, όπου οι, οι συνθήκες για τους νέους εκεί είναι τέτοιες που κάποιοι από αυτούς ε, θα μπορούσαν να πούν ότι αυτό το επίπεδο οργανωμένης βίας ε, και η ανικανότητα του κράτους να τους προστατεύσει είναι επαρκή στοιχεία για να θεωρηθούν πρόσφυγες και να χρήσουν διεθνούς προστασία η αξιοπρεπή μεταχείριση ενός παράτυπου μετανάστη ε, δεν μπορεί να θεωρηθεί κίνητρο στο να έρθουν και άλλοι. Το ξαναλέω. Το λέω αυτό επί της βάσης ότι σε έναν άλλον τομέα όπου έχω εργαστεί στο παρελθόν, ε, στο ποινικό δίκαιο, η ιδέα του αποτρεπτικού χαρακτήρα πρέπει πάντα να εξετάζεται πολύ προσεκτικά. Η τιμωρία συχνά θεωρείται ως ένα αποτρεπτικό στοιχείο. Είναι δηλαδή ε, μια τιμωρία όχι μόνο για τη δικαιοσύνη, για λόγους δικαιοσύνης, αλλά και διότι θεωρούμε ότι αυτό θα αποτρέψει ε, τέτοιες συμπεριφορές. Σίγουρα η φυλάκιση ε, αποτρέπει το συγκεκριμένο άτομο, ο οποίο είναι στη φυλακή και δεν μπορεί πλέον να δράσει παράνομα. Το κατά πόσο όμως αυτό έχει αποτρεπτικό αποτέλεσμα σε άλλους, είναι πολύ πιο προβληματική ε, συζήτηση, πολύ πιο δύσκολη. Είναι κάτι το οποίο αφιζητούν ιδιαίτερα όσοι είναι κατά της θανατικής ποινής και κατά τη γνώμη μου καλά κάνουν και το αμφισβητούν. Ε, βασιζόμαστε στην υπόθεση ότι όλοι είναι στην ίδια κατάσταση. Στον τομέα της μετανάστευσης αυτό, αυτή η υπόθεση είναι εξαιρετικά έολη θα πρέπει δηλαδή το ίδιο άτομο υπό τις συνθήκες να πούμε ότι θα αντιδράσει με τον ίδιο τρόπο. Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η απόφαση που παίρνει κάποιος για να φύγει από τη χώρα του ε, έχει να κάνει με πάρα πολλούς παράγοντες, πολύ προσωπικούς παράγοντες ε, και έχουν να κάνουν κυρίως με την ανάγκη του να φύγει κάποιος από εκεί που είναι πολύ περισσότερο από ότι ε, κα, την, ε, το κατά πόσο προσελκύει ο τόπος προορισμού και ακόμα και αυτά τα κίνητρα προσέλκυσης έχουν να κάνουν με οικογενειακούς παράγοντες, με γλωσσικούς, πολιτιστικούς παράγοντες και όχι το κατά πόσο ε, υπάρχει κάποια νομοθεσία εκεί η οποία θα του είναι ευνοϊκή. Ε, νομίζω πως είναι λάθος αυτό το επιχείρημα. για το κλίμα, για την κλιμα... τους κλιματικούς μετανάστες. Είπα ότι ε, προφανώς και θα αναγνωριστεί ο αυξανόμενος αριθμός περιβαλλοντικών παραγόντων ε, ως παράγοντες ε, μετανάστευσης. Και αυτό θα αυξηθεί τις επόμενες δεκαετίες. Κατά πόσο τώρα θα φτάσουμε σε ένα σημείο όπου μέσω μιας άλλης σύμβασης, μιας άλλης συνθήκης, μέσω ενός πρωτοκόλου στην σύμβαση για τους πρόσφυγες, τα κράτη-μέλη των ΗΕ θα είναι διατεθειμένα να διαπραγματευτούν μια σύμβαση που θα δίνει ε, συγκεκριμένη νομική διεθνή προστασία προς τους ε, κλιματικούς πρόσφυγες μετανάστες. Ε, δεν είμαστε ακόμα, δεν έχουμε φτάσει εκεί. Σε αυτή τη φάση το καλύτερο είναι να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τους μετανάστες ε, σε ευάλωτη κατάσταση. Ε, αυτό περιλαμβάνει και τους περιβαλλοντικούς μετανάστες και άλλους πολλούς. Uh, ε, ευχαριστώ που απαντήσατε σε όλες τις ερωτήσεις και τα σχόλια. Η Λίντα Μάκαβαν για να κλείσει αυτή η κοινή συνεδρία. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Λουίζ Άρμπορ είχατε την καλοσύνη να μας δεχθείτε πέρυσι τον Ιούλιο που είχαμε μεταβεί με αντιπροσωπεία της Επιτροπής μας στη Νέα Υόρκη. Πραγματικά τηρήσατε στο ακέραιο την υπόσχεσή σας να είστε σε επαφή με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πολύ σημαντικό. Καλά κάνετε και μας θυμίζετε ότι οι χώρες μας έχουν δικαιώματα αλλά έχουν και ευθύνες και υποχρεώσεις. Και εμείς που έχουμε δημόσιο λόγο θα πρέπει να το τονίζουμε αυτό και ξέρουμε πολύ συχνά χρησιμοποιείται ε, ως επιχείρημα η μετανάστευση για προεκλογικές σκοπιμότητες και ε, λόγους. Θέλω, ε, σας ευχαριστώ που ήρθατε. Θέλω να θυμίσω στους συναδέλφους Επιτροπής Ανάπτυξης ότι θα συνεδριάσουμε σε άλλη αίθουσα 3Ε2. Η επιτροπη ΔΕΒΕ Ντέβε συνεδριάζει 3Ε2 όπου θα έρθει να μας μιλήσει ένας επικεφαλής Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας. Ευχαριστώ και ξαναδίνω το λόγο στον Ντέιβιτ και την Επιτροπή Εξωτερικών.